Σύμφωνα με τον κώδικα διοντολογία των ε, βουλευτών σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και συγκρούσεων συμφερόντων, στι 5 Απριλίου αποφάσισα να ορίσω την κυρία Ντανούτα Χούμπνερ, την κυρία Μάντελβο, τον κύριο Σαγιάντ Καρύμ τον κύριο Ζαμαρί Καβαντά και τον κύριο Γύρι Μαστάλκα ω μέλη τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τον Κώδικα Διοντολογία των ε, Βουλευτών και επίση την κυρία Χέιντι Χάουταλα, την κυρία Λάουρα Φεράρα, τον κύριο Γκέρολ Φάνεμα ως μέλη αναπληρωματικά της Συμβουλευτικής αυτής Επιτροπής.